και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το χρόνο γιατί έχουμε καθυστέρηση λιγάκι. Θα πρέπει να συζητήσουμε, να συζητήσουμε την κατάσταση των Ροχίνγκα, τη ε, μουσουλμανική αυτή μειονότητα στην ε, Μιανμά, Θα δώσω καταρχήν το λόγο στου συντάκτε των ψηφισμάτων, πρώτα τον κύριο Ντεμέσμακερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρία Πρόεδρε, έχουμε κάτοχο βραβείου Ζαχάροφ, ήρωα ε, της σύγχρονης εποχής, την Αούν Σανσουκή που το 2011 ε, κερδίζει για τη Δημοκρατία και τη χώρα της το Μιανμάρ ε, και παρόλα αυτά ε, βλέπουμε κάποιες ε, καταστάσεις ε, για τους Ροχίνγκια, την μειονότητα αυτή που από το 82 την αρχή της στρατιωτικής δικτατορίας στο Μιανμάρια είναι απάτριδες, ανηθαγενείς όπως λέει το ψήφισμα. Πολλοί έχουν διαφύγει σε άλλες χώρες, αλλά πολλοί ζουν σε καταβλισμούς, τους κακομεταχειρίζονται, δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, τρόφιμα λόγω αυτής της ανελαίτης πολιτικής πρόκειται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει και η ΕΕΔ να θέσει το ζήτημα στο ύψιστο δυνατό επίπεδο και να καλέσει τη Μιανμάρ και άλλες χώρες και στο υψηλότερο επίπεδο ε, να το θέσουμε το θέμα με την ΜΑΜΑΡ και τις άλλες ασιατικές, μάλλον τις χώρες του ΑΣΕΑΝ ώστε και η πατιαρμοστία να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την κατάσταση του καταβλισμού των και Ευχαριστώ λέει πρόεδρος η κυρία Χάουταλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα καλύτερα νέα της τελευταίας χρονιάς στον τομέα της διεθνούς πολιτικής ήταν ότι από στρατιωτική δικτατορία πέρασε σε ένα διαφορετικό καθεστώς ε, η χώρα του Μιανμάρ. Σίγουρα ε, περιμένουμε, παρότι αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, ε, περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη και την πρόσφατη έκθεση του προσώπων των ΗΠΑ για τους Ροχίνγκια και τις άλλες μειονότητες της Βυρμανίας. Κάθε μορφή διάκριση πρέπει να εξαλειφθεί. Η Αούν Σανξουκή βλέπουμε ότι αρχίζει να διαφέρει και για τους Ροχίνγκια πλέον. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω. Το ζήτημα αυτό φρενάρει και την ανάπτυξη του Μιανμάρ. Τελειώντας να αναφέρω ένα πράγμα μόνο. Όλα τα δυτικά κράτη και η Κίνα θέλουν να έχουν εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές με το Μιάνμα. Επομένως θα πρέπει η κυβέρνηση της χώρας ε, να ε, βοηθήσει να υπάρξουν υπεύθυνε εξαγωγές των ε, φυσικών πόρων και να υπάρχει μια ανοιχτή στάση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και Σκοράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σε αυτή την περίπτωση συζητάμε εκ την ε, μειονότητα των Ροχίνγκα με, σε, ένα χρόνο, με ένα χρόνο την τελευταία φορά. Δυστυχώς οι συνθήκε διαβίωση του λαού των Ροχίνγκα δεν άλλαξαν καθόλου. Έχουν μάλιστα επιδεινωθεί και παίρνουν τη μορφή μια γενοκτονίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Μιαμάρα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωση σίγουρα θα μπορούσε να είναι ισχυρότερο ε, στο διάλογο με την Μιανμάρ αλλά και με τις γειτονικέ χώρες που απορρίπτουν ε, που μάλλον που αποθούν όταν από την άλλη πλευρά γίνονται διαρκώς συλλήψεις. Έχει γίνει καλή δουλειά από την DG όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Φτάσαν περίπου 70 εκατομμύρια από το 2010 μέχρι σήμερα και πρέπει να πιέσουμε την νέα κυβέρνηση όπως έλεγαν και πριν κάποιοι ομιλητέ, για να προσπαθήσουμε ακριβώς να αλλάξουμε το ρυθμό και να προστατεύσουμε αυτή την μειονότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλαμ τώρα. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Εμεί εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία σας σε αυτή τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί αυτό καταδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η μειονότητα των Ροχίνγκιας είναι ένα ειδικό θέμα, το οποίο δεν έχει γίνει πλήρως αναγνωριστό ή κατανοητό. Για πολλά χρόνια όχι μόνο αντιμετώπισαν διακρίσεις, αλλά βρίσκονται σε υπαρξιακό κίνδυνο επιβίωσης. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση ότι μια ολόκληρη εθνοτική ομάδα δεν αναγνωρίζεται σε μια χώρα όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς. Δεν αναγνωρίζονται ως πολίτες της Μιανμάρ και θεωρούνται ανεπιθύμητοι εκεί. Η νέα κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει αποφασίσει να προχωρήσει με προτεραιότητα στην εθνική συμφιλίωση. Γι' αυτό τους ζητούμε να δώσουν ασφάλεια στους Ροχίνγκα και να σταματήσουν την ατιμορρησία και να τους δώσουν προστασία και ηθαγένεια στην Μιανμάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο ο συντάκτης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση νομίζω πως είναι αρκετά σαφής και προφανής. Δεν χρειάζεται να επαναρχόμαστε. Το Πρέπει να δώσουμε ε, μία όθηση σε αυτή την κατάσταση, να κάτι να γίνει. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα των Ροίγκα που ζουν σε χείριστες συνθήκες και πολλοί φεύγουν από τα σύνορα προς τον Μπαγκλαντές. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ ορισμένου καταβλισμούς στα σύνορα ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ και εκεί πραγματικά ε, υπάρχουν εκκρεμή προβλήματα. Πρέπει να γίνουν ένα-δύο πράγματα, πιστεύω. Καταρχάς να πιέσουμε τη σημερινή σημερινή κυβέρνηση της Μιανμάρ που είναι σε φάση δημοκρατικής μετάβασης και να πούμε πως είναι απαράδεκτες οι σημερινές συνθήκες διαβίωσης των Ροίγκα. Είναι σαν απαρτχάιτ. Και το δεύτερο είναι αν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί για να φτιάξει ένα νέο μνημόνιο ανάμεσα στην Μιανμάρ και τη Ταϊλάνδη για να λυθεί και το πρόβλημα των, πληθυσμών, των πληθυσμών που βρίσκονται στην Ταϊλάνδη απομακρυσμένοι και πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάτε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Μογκερίνη, οι Ροχίνγκα έχουν ε, υποφέρει από βίαιη καταπίεση και διακρίσεις φεύγουν από την Μιαμάρ και πολλοί χάνονται στο δρόμο. Παιδιά και μητέρες χάνονται, πεθαίνουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Τα παιδιά δεν καταχωρούνται στα μετρώα όταν γεννιούνται, δεν μπορούν να πάνε σχολείο, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό πρέπει να πάψει. Για πρώτη φορά σε 50 χρόνια η Μιανμάρ πέρασε στην πρώτη μη στρατιωτική πρόεδρο του, της χώρας από το 1962 είναι μια νέα δυνατότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια. Η Μιανμά πρέπει να αλλάξει. Οι διαμάχες πρέπει να λυθούν μέσω διαπραγματεύσεων. Η, η μειονότητα Ροχίνγκα θα πρέπει να λάβει την ηθαγένεια και οι, οι ε, τοπικές νομοθεσίες εναντίον της να καταργηθούν. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα μέσω project, μέσω συμφωνιών όπως με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Βεζιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά μιλάμε για τη μειονότητα Ροχίνγκια που διώκεται από τι πιο διωκόμενε. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι που δεν έχουν ηθαγένεια, που του κυνηγούν παντού. Η Ροχίνγκια είναι μια λέξη που στη Βερμανία δεν πρέπει καν να προφέρεται. Η Αούν Σανσουκή πρόσφατα θύμισε στους πρέσβεις και υπευθύνους ε, το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Καλή η νίκη του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία. Αλλά όλα είναι εύθραυστα. Οκτώ μήνες μετά τις εκλογές συνεχίζεται η καταστολή. Πράγματι, τεράστια επρόκληση νομική, αρχιτεκτονική βασίζεται σε διακρίσεις, ε, στις ε, εθνοκοστρισκευτικές διαφορές πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπάρχουν τέσσερις νόμοι προστασίας ε, της φυλής ε, από το 1975 και άλλοι νόμοι που πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχει επίσης έκρηξη βίας, ισλαμόφοβη, λόγω του ριζοσπαστικού βουδισμού που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δύο τεμένοι μέσα σε μια εβδομάδα καταστρέφηκαν στο βορρά και στο κέντρο της χώρας. Ελπίζουμε η συμβολική διάσκεψη του Πανκ Λόγκ, αν βέβαια συμμετέχουν όλοι, να βοηθήσει στην ειρήνευση στη χώρα πέραν και του κατεπίου του ζητήματος των Ροχίνγκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να μην ε, υπερβαίνετε το χρόνο σας, αλλά και να μην μιλάτε τρομερά γρήγορα, γιατί δεν είναι δυνατόν να σας ε, διερμηνεύσουν. Κύριε Σβόποντα, για ένα λεπτό ως πρώτος από τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η Μιανμάρ έχει μια κυβέρνηση της οποίας ηγείται μια βραβευμένη με βραβείο Σαχάρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα δεν είναι ότι έχουμε κάνει τα απαραίτητα. Δυστυχώς η κατάσταση των Ροχίνγκα στην Μιανμάρ δεν έχει βελτιωθεί, μάλλον χειροτερεύει. Ακόμα δεν έχουν ηθαγένεια, υπάρχει ανακτικότητα της γενοκτονίας εναντίον τους από τους βουδιστές. Αντιμετωπίζουν λοιπόν υπαξιακό κίνδυνο. Δεν επιτρέπεται να έχουν πάνω από δύο παιδιά για να μην ευχεί δημογραφική ανάπτυξη η ομάδα τους. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Μιανμάρ. Οι λήπτες αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πούν σαφώς ότι μια τέτοια μεταχείριση μιας εθνοτικής ομάδας είναι απόλυτα απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή με κανένα τρόπο η γενοκτονία εναντίον δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η κυρία Άννα Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τη κυρία Μογκερίνη στη συζήτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση στη Μιανμάρ που ήταν αποτέλεσμα δημοκρατικών εκλογών που είχα και εγώ την τιμή να παρακολουθήσω ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σίγουρα θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία της δημοκρατίας και θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αποτροπή των διακρίσεων και των διώξεων κατά των Ροίγκα και άλλων εθνοτικών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό και μόνο μπορεί να υπάρξει εθνική συμφιλίωση. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει και κύρωση και ποινικέ κυρώσει εναντίον όλων των ηγετών των βουδιστών που κάνουν βίες ενέργειες κατά τον Ροχίγκα. Η άγξουση έχει μεγάλη ευθύνη ως ε, μέλος της κυβέρνησης στη Μιανμά και ως εμβληματική φυσιογνωμία για τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στη χώρα της αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να ζητήσει δημόσια την προστασία των Ροχίνγκα και θα πρέπει να διευκολύνει και την παρουσία των διεθνών φορέων και θα πρέπει να προτείνει τις απαραίτητες συνταγματικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα πρέπει να ασκήσει πίεση, αλλά θα πρέπει να ασκήσει και πίεση στις άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών που έχουν προβλήματα με τους Ρόγιγκα και δεν σέβονται την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Ο κύριος Μαριάς. Μαριάς, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει με τους άλλους συναδέλφους. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιαμάρ είναι συχνό φαινόμενο, με τις διώξεις και τη βία κατά της μειονότητας των Ροχίγκα να εντείνονται διαρκώς. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας των Ροχίγκα και των τόπων λατρείας τους οι μαζικές συλλήψεις η αυθαίρετη φυλάκιση και οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των αρχών της μιανμάρ απέναντι σε αυτή την μειονότητα. πάνω από 130.000 εκτοπισμένοι ροχίγκα παραμένουν σε στρατόπεδα σε άλλες περιοχές ενώ οι αρχές της μιανμάρ έχουν καταστήσει ανεπαρκή την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές παράλληλα εκτιμάται ότι 10.000 χιλιάδες έχουν τραπεί σε φυγή διαθαλάσσης για να γλιτώσουν τον διωγμό και 1.700 κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες σε κέντρα κράτησης για πρόσφυγες. είναι αναγκαίο επομένως οι αρχές της μιανμάρ να επιτρέψουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθεια σε όλες τις περιοχές της χώρας και να δράσει άμεσα η ευρωπαϊκή ένωση για τη στήριξη των δικαιωμάτων των ροχίνγκα. ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιο Ιππίντου. Για ένα λεπτό. Η τραγωδία των Ροίγκα στη Μιανμάρ έχει τόσες που είναι τόσο πολυδιάστατη που εγγύζει τη βαθύτερη μας ε, ηθική, ηθική και πολιτική συνείδηση. Αυτή η μειοψηφία διώκεται από τις αρχές της ε, Μιανμάρ που δεν τους αναγνωρίζουν καν ως πολίτες της χώρας. Υποχρεώνονται λοιπόν να εγκαταλείψουν τη χώρα ε, υπό πολύ ε, επισφαλείς συνθήκες. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά προσπαθούν ε, να φύγουν μέσω από σκοτεινά δίκτυα διακινητών ανθρώπων, περνάνε τα βουνά χωρίς νερό και μάλιστα πολλές φορές τους δολοφονούν κιόλας η Ισλαμοφοβία όλο ένα και εντονότερη στην Ευρώπη είναι καλό οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να πείσουν την κυβέρνηση της Μιανμάρ ότι υπάρχουν περισσότερα πλονεκτήματα στο σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μειονότητας μάλλον των Ροχίνγκα παρά με την παραβίασή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ταραμπέλα, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπη, αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο πριν ένα χρόνο ξανασχοληθήκαμε εδώ με την καταστροφική κατάσταση των Ροίγκα στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Μιανμάρ. Αυτό ο Γολγοθά που, ε, που ζει ένα εκατομμύριο κόσμο είναι φρικτός. εκπρόσωπος των, ε, του ΟΗΕ, εκπρόσωπος μάλλον του ΟΗΕ που ήταν στην ε, Μιανμάρ πριν από λίγο δεν διαπίστωσε καμία πρόοδο παρά τη δημοκρατική μετάβαση στη χώρα. Ο ΟΗΕ μάλιστα δημοσίευσε ιδιαίτερα αυστηρή έκθεση ε, έναντι της Μιανμάρ και καταγράφονται εκεί διώξεις στις οποίες υπόκειται ο λαός των Ροίγκα θα πρέπει να αναγνωριστεί επιτέλους ένα πραγματικό καθεστώς σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί η Μιανμάρ δεν τους αναγνωρίζει ε, ηθαγένεια ούτε βικότητα ε, άρα είναι ε, απάτριδες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους και επίσης η πρωτοβουλία του κύριου Πανζέρη για την επιστροφή των εκπατρισμένων από την Ταϊλάνδη προς την Μιανμάρα. Ευχαριστώ. Και το... Περνάμε στη δικασία προσέγγισης προσέγγισης του Προέδρου. 2 έχουν στήσει το λόγο. Πόσπισιλ καταρχά. Κύριε Πόσπισιλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πριν από λίγους μήνες ε, είχα ασκήσει κριτική στην κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σε καμία περίπτωση. Στηρίζω λοιπόν ό,τι είπαν οι προλαλήσαντες, ε, οι ροχίγκας ε, χάνουν την ηθαγένειά τους. Δεν έχουν ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι άκρος λυπηρή αυτή η κατάσταση διότι έχουμε βραβευτεί σαν βραβείο Ζαχάροφ ε, στην κυβέρνηση, η οποία όμως δεν έχει κάνει κάτι για να βελτιώσει την κατάσταση της μουσουλμανικής αυτής μειονότητας. Αυτό είναι άκρος λυπηρό και εξού και χρειαζόμαστε τώρα ένα νέο ψήφισμα με το οποίο ζητούμε τη δημοκρατική κυβέρνηση στην οποία συμπεριλαμβάνεται την κυρία Σουκή, να κάνει κάτι για αυτή την φρικτή κατάσταση. Έλληνες δεν μπορεί να γίνεται λόγος για δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, πρόεδρος. Ευχαριστώ παρακαλώ. Υπάρχει πολύ θόρυβο στην αίθουσα. Σας παρακαλώ να κάθεστε ησύχως. Κύριε Κού, είστε ο τελευταίο ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, έχουμε παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον την δημοκρατική μετάβαση που έχει γίνει στη Μιανμά. Ελπίζουμε ότι αυτή η αλλαγή θα βελτιώσει την κατάσταση όλων των πολιτών στην χώρα αυτή αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση μειονοτήτων όπως η Ροχίνγκια. Η καταδίωξη των Ροχίνγκα έχει μακρά ιστορία στην Μιανμάρ. Τα τελευταία χρόνια είδαμε κύματα προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων από την κοινότητα των Ροχίνγκια και πολλές ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και διώξεις καθώς και διακρίσεις εναντίον τους. Αυτή η ομοιονότητα είναι μία από τις πιο καταδιωκόμενες μειονότητες σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση λοιπόν της Μιανμάρ θα πρέπει να δείξει σεβασμό για τα δικαίωματα όλων αυτών των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτή τη μειονότητα και αυτό αφορά και τις άλλες χώρες της γειτονικές περιοχής. Οι χώρες που έχουν μεγάλο αριθμό προσφύγων Ροχίνγκα θα πρέπει να εξασφαλίσουν την προστασία τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν αυτό το μακρό αφήγημα σε σχέση με τους Ροχίνγκα. Θα ήθελα να ζητήσουμε την κυρία Μογκερίνη να μα απαντήσει σε όλα αυτά που είπαν οι βουλευτές. Σας παρακαλώ να έχουμε λίγη ησυχία στην για να ακούσουμε την υπάτη εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται ούτε να με ακούσετε ούτε και να είστε ε, σιωπηλοί. Απλά να κάθεστε σιγά σιγά. Όσοι λάβατε το λόγο, αξιότιμοι βουλευτέ, ε, σε αυτή τη συζήτηση γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαδραματίζει ένα σημαντικό ειδικό ρόλο σε ό,τι αφορά Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε διεθνεί παρατηρητέ ε, στη Διεθνή Συμφωνία Εκεχηρία και αυτό μα δίνει μια ειδική ευθύνη και ένα ιδιαίτερο ρόλο όπου περιλαμβάνονται διάφορα αισθήματα όπως αναφέρατε. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ιστορική ευκαιρία με τη νέα κυβέρνηση. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την κυβέρνηση σε διάφορους τομείς, μείωση της στόχιας, μετανάστευση, και βέβαια και για την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια και θα συναντηθώ ε, με την πρόεδρο του Μιανμάρ ε, στο επόμενο, στην επόμενη διάσκεψη της κορυφής ε, των χωρών Ασιαν και με άλλους ηγέτες βέβαια της περιοχής για να επαναλάβουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντί τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή Ρακίνα, την πολιτεία αυτή στην οποία κυρίως διαμένουν οι Ροχίνγκια, Είχα συναντηθεί και με τον Τέο Υπουργό πέρυσι. Υπάρχει και ο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση Μιανμάρ και στο πλαίσιο αυτού, ο ειδικό εκπρόσωπο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριο Λαμπρινίδη και πάλι που είναι και μαζί μα σήμερα, επισκέφθηκε ε, την πολιτεία Ρακίνα για να εκτιμήσει την κατάσταση και να ζητήσει μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε επίσης έχουμε καταθέσει ορισμένα ψηφίσματα για ε, την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει στην περίπτωση των Ροχίνγκια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ανέφεραν το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο υπήρξε ένας βασικός πολιτικός συνομιλητής αλλά και βασικός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Ροχίνγκια. Το 2016 πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ που θα πει 68% ε, του ανθρωπιστικού προεπολισμού για ε, το Μιανμάρ έχουν δοθεί για την πολιτεία αυτή ε, στην οποία διαμένουν Ροχίνγκια για να υποφεληθούν οι άνθρωποι αυτοί. Παρέχουμε υποστήριξη ιδίω ε, στην ε, βοήθεια για την εκπαίδευση των παιδιών και την εκρίζωση της φτώχειας σε αυτό το τμήμα της χώρας. Η κυβέρνηση η κυβέρνηση της Μιανμάρ αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και εμείς φροντίζουμε να παραμένουν προσιλωμένοι στην πρόθεσή τους να βελτιώσουν την κατάσταση. Η Αουν Σαντσουκή κάνει και αυτή ε, βήματα για να βρει βιώσιμες λύσεις για τις δεκοινότητες, ηγείται μιας επιτροπής, η οποία έχει ως στόχο να φέρει η ειρήνη, η σταθερότητα, ανάπτυξη στην περιοχή. Υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης θαγένειας, ξεκίνησε αρχές Ιουνίου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, των Ροχίνγκια αλλά και άλλων μειονοτήτων. Σίγουρα γι' αυτό χρειάζεται χρόνος, εξού και χρειάζεται και τη συνεχή μας υποστήριξη αυτή η προσπάθεια. Όπως είπα λοιπόν εντείνουμε ε, τι σχέσει μας με τη Μιανμάρ για να ε, επιλύσουμε τα προβλήματα σύμφωνα και με τη στρατηγική και την κοινή ανακοίνωση που εγκρίναμε στις αρχές Ιουνίου. Όπω και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να ξεκινήσει ένα ε, αξιόπιστο πρόγραμμα δράσης κατά των διακρίσεων και για αλληλέγγυα και για όλους ε, ένταξη. Ελπίζουμε να υπάρξει μια πραγματική συμφιλίωση στη χώρα. Ολοκληρώνοντα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία ειρήνευση και ε, συμφιλίωση, ιστορική διαδικασία στη Μιανμάρ, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλε τι αρνητικέ θρησκευτικέ ομάδε και προ αυτό εργαζόμαστε και εμεί, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ιπατέκ εκπρόσωπε ζητώ συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να επιβάλλω ησυχία στο ημικύκλιο. Έχουμε 7 ψηφίσματα, 7 προτάσεις ψηφίσματος. Και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση.